Επιτέλους, μετά από 10 χρόνια συζητήσεων, βρισκόμαστε εδώ, μετά από πολλά εμπόδια, πολλές τροφές. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση Καπούρης για την ε, υπομονή τη και τον πρέσβη τη Σιγκαπούρη για την καλή συνεργασία του. Επίση, θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν και την Γενική Διεύθυνση Trade για μια συμφωνία την οποία μπορούμε πιστεύω να στηρίξουμε. Επίση, θα ήθελα να ευχαριστήσω του και ηγητέ για την πολύ καλή συνεργασία. Κάποιοι μπορεί να είναι ακόμα σκεπτικοί, στες, ε, τι δεν είναι καλό για αυτή, ε, σε σχέση με αυτή τη συμφωνία. Αυτή η συμφωνία βασίζεται στη συμφωνίε με τον Καναδά και την Ιαπωνία. Στέλνει το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προσιλωμένη σε ένα σύστημα εμπορίου που θα βασίζεται σε κανόνε, ενώ ο Ντόναλτ Τραμπ θέλει να στήσει τείχου και τείχη. Εμεί του καταργούμε και δημιουργούμε ζώνες ελεύθερων συναλλαγών. Η Σιγκαπούρη είναι ένα ασφαλές καταφύγιο για ε, το ευρωπαϊκό εμπόριο και τις επενδύσεις και τι, και τι καταφύγιο, ένα σημαντικό, μια σημαντική αγορά, μια χώρα που είναι προσιλωμένη στο κράτος δικαίου, ε, με ένα από τα υψηλότερα κατά κεφαλή εισοδήματα στον κόσμο. Πάνω από 10.000 ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν ε, την βάση τους εκεί. Και πολλές από αυτές, ε, με εργαλείο αυτή τη συμφωνία, θέλουν να διευρύνουν τι δραστηριότητε τους στη Σιγκαπούρη μέσω, των, μέσω εταιρικών σχέσεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Είναι και στρατηγική σημασία χώρα η Σιγκαπούρη για να έχουμε πρόσβαση στην ε, ασιατική περιοχή, στην περιοχή αυτή της Ασίας, η οποία αναπτύσσεται με ταχύτητα τους ρυθμούς. Ένα μεγάλο ποσοστό των εξαγωγών μας προς την περιοχή αυτή περνούν ε, από τη Σιγκαπούρη. Και αν δεν κάνουμε τίποτα, δεδομένου ότι η Σιγκαπούρη έχει ήδη εταιρική σχέση με τις χώρες του Ειρηνικού, θα μείνουμε πίσω. Από οικονομικής πλευράς είναι λοιπόν αμοιβαία ωφέλιμη αυτή η συμφωνία. Όμως επιπλέον των εμπορικών ωφελών θα μπορούσα να πω ότι η συμφωνία αυτή αντικατοπτρίζει σαφώς και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και τις θέσεις του Κοινοβουλίου που έχουν επαναληφθεί επανειλημμένως στο παρελθόν. Για παράδειγμα, τίποτα σε αυτή τη συμφωνία ε, δεν θα εμποδίσει την εφαρμογή της αρχής προφύλαξης προκειμένου κυβερνήσει να μοθετούν οι όφελο των πολιτών τους. Ε, προστατεύονται οι δημόσιες υπηρεσίες, ε, οι εισαγωγέ θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα, ευρωπαϊκέ προδιαγραφέ, προδιαγραφές, ε, προσήλωση στην, προσήλωση, ε, στην προστασία του περιβάλλοντος, της τη γεωργίας και ε, προϋποθετήθεται η σύναψη άλλων διεθνών συμφωνιών όπως η Συμφωνία του Παρισιού. Επίσης αναλαμβάνεται από τη Σιγκαπούρη η υποχρέωση να υπογράψει τις τρεις συμφωνίες του ΑΕΛΟ, της Διεθνούς Οργανωσής Εργασίας, που δεν έχει υπογράψει ακόμα. Ε, επίσης, ε, ε, ε αναλαμβάνουν την ευθύνη να δημιουργηθεί μια ομάδα, διαϋπουργική ομάδα, προκειμένου να εφαρμοστούν αυτές οι συμφωνίες σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών. Είναι η πιο προοδευτική επενδυτική συμφωνία που έχουμε διαπραγματευτεί μέχρι τώρα και θα πρέπει να αποτελέσει μοντέλο για το μέλλον. Θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν και την όλη ομάδα της ε, για το ρόλο του στη διαπραγμάτευση. Ε, προβλέπεται ένα μόνιμο ε, επενδυτικό δικαστήριο, έναν διοντολογικό κώδικα για τους δικαστές, ένα μηχανισμό έφεσης και ε, τη χρήση του πολυμερούς Διεθνούς Δικαστηρίου των Διαφορών. Αντικαθιστά τις 13 διμερείς σχέσεις προστασία των επενδύσεων που έχουν αυτή τη στιγμή κράτη-μέλη με τη Σιγκαπούρη. Υπάρχει μία δυναμία σε αυτή τη συμφωνία που θα πρέπει να καλυφθεί στις μελλοντικές συμφωνίες. Τους δίνει στους επενδυτές δικαιώματα, αλλά όχι υποχρεώσεις με αυτή την επιφύλαξη μπορώ και τις δύο συμφωνίες να τις ε, συστήσω προς ψήφιση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μαρτίν, λέει ο πρόεδρος. Έχω ένα αίτημα, έχουμε καθυστερήσει, είμαστε καθυστερημένοι για κατά 15 λεπτά. Παρακαλώ πολύ, ας παραμείνουμε ο καθένας στο χρόνο που του δίδεται για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση πριν τα μεσάνυχτα. Οπότε δεν θα κάνω δεχτέ τι μπλε κάρτε. Ο άλλος εισηγητή, ο κ. Λόπεθ, Στουρι Σουάιτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο Ντέβιτ Μάρτιν. Θέλω και εγώ να συγχαρώ, να ευχαριστήσω τον πρέσβη τη Σιγκαπούρη. Μα βοήθησε πάρα πολύ ε, στην επεξεργασία αυτών των νομοδοτήσεων, των εκθέσεων. Ε, μας έδωσε με διαφανή τρόπο πολλές πληροφορίες για τη Σιγκαπούρη. 15 χρόνια έχουν περάσει από τότε που ξεκίνησε, που μάλλον το Συμβούλιο ζήτησε από την Κομισιόν να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Εδώ τελειώνει η διαδικασία αυτή. Αύριο θα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα με την ψηφοφορία. Ε, προκειμένου να συμφωνήσουμε με το πλαίσιο συνεργασίας και τις συμφωνίες προστασίας των επενδύσεων ε, των επενδυτών. Μία ακόμα φορά στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα για την δέσμευση της Ένωσης στην πολυμερή διεθνή συνεργασία σε θέματα εμπορίου, αντίθετα με άλλου. Σε αυτή τη στιγμή αυτή η πολυμερή προσέγγιση τίθεται υπό αμφισβήτηση. Εμείς επιμένουμε στη διεθνή συνεργασία. Αυτή η συμφωνία προσπαθεί να θεσμοθετήσει σχέσει οι οποίες υπάρχουν εδώ και πολλές δεκαετίες βασίζονται σε μακρά ιστορία φιλίας και οικονομικούς, ε, κοινωνικούς και πολιτικούς δεσμούς. Ε, θα αποτελέσει ένα νομικό πλαίσιο για την συνεργασία μεταξύ Συγκαπού και Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Στόχος είναι η συνεργασία σε θέματα δικαιοσύνη, ασφάλεια, κλιματική αλλαγή και ανάπτυξη μεταξύ άλλων. Ε, πράγματα τα στα οποία δίνουν ιδιαίτερη σημασία οι πολίτες μας. Η Σιγκαπούρη είναι σημαντικός παράγοντας για να εξασφαλιστεί η περιφερειακή ισορροπία στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού. Κάτι που είναι σημαντικό για την Ευρώπη, για τις επιχειρήσεις μας και για τους Ευρωπαίους πολίτες. Η Σιγκαπούρη είναι η πόρτα εισόδου στην ασιατική αγορά και μια πλατφόρμα για τι ε, ευρωπαϊκέ επιχειρήσει. Βρίσκεται στρατηγικά τοποθετημένη κοντά στην Ιαπωνία, την Κίνα και άλλε οικονομίε, σημαντικέ οικονομίε τη Η συμφωνία αυτή θα δώσει μεγαλύτερη ασφάλεια στου Ευρωπαίου επενδυτέ. Να υπογραμμίσω ότι στο πλαίσιο αυτή τη συμφωνία θα δημιουργηθεί μια μόνιμη μεικτή επιτροπή με αντιπροσώπους των δύο πλευρών σε υψηλό επίπεδο, έτσι ώστε καθημερινά να εργάζονται προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι συνεργασία. Θα Είμαστε σημαντικοί συνομιλητέ σε θέματα που θα έχουν σχέση με την διεθνή ασφάλεια, την συνεργασία σε τεχνολογικό, ερευνητικό επίπεδο, το περιβάλλον, του φυσικού πόρου και τι μεταφορέ, ιδιαίτερα τι θαλάσσιε και αέριε μεταφορέ. Θα συνεργαστούμε σε θέματα ε, πληροφορία ε, ε, και ανταλλαγή πληροφοριών οι επιχειρήσεις μας αυτή τη ε, στιγμή, για παράδειγμα, χάνουν πολλά εκατομμύρια από επί, κυβερνοεπιθέσεις, τις οποίες θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη συνεργασία. Ε, πολιστικές ανταλλαγές ήδη υπάρχουν, θα τις διευρύνουμε. Προγράμματα ε, όπως το Μούντι και το Εράσμους ε, ε, θα διευρυθούν και θα εφαρμοστούν και για τη Σιγκαπούρη. Η Σιγκαπούρη μπορεί να γίνει πλατφόρμα για τους νέους μας προς τις χώρες της Ασίας. Επίση, είναι σημαντική για τη συνολική παγκόσμια ασφάλιση και την ασφάλεια και την καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Η συνεργασία είναι ο μόνο τρόπο να καταπολεμήσουμε αυτή τη μάστιγα. Χρειαζόμαστε γέφυρε συνεργασία με τι άλλε χώρε, ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων. Ε, ε μείωση της χρηματοδότησης ε, και γενικότερη καταπολέμηση της τρομοκρατίας συμφωνία αυτή θα είναι πολύ καλή λοιπόν και για τους επιχειρηματές και για τις επιχειρήσεις ε, για να δημιουργήσουν σχέσεις όχι μόνο με τη Σιγκαπούρη αλλά και με άλλους χώρε τη Ασία. Πάνω από 10.000 ευρωπαϊκέ επιχειρήσει και επιχειρηματίε βρίσκονται ήδη στη Σιγκαπούρη, την χρησιμοποιούν ω κέντρο για να εξυπηρετήσουν όλη την περιοχή του Ειρηνικού. Ένα μόνιμο νομικό πλαίσιο θα αποτελέσει ακρογωνίο λίθο τη συνεργασία μα ε, και θα δώσει νομική ασφάλεια στι επιχειρήσει μα. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγουμε καινούριε ευκαιρίε εμπορίου, προάγουμε τι επενδύσει, την ανάπτυξη και τη διεύρυνσή του. Κάθε φορά που οι πολίτε μα μπορούν να αναπτύσσουν τι ιδέε του και τα σχέδιά τους με τρόπο ασφαλή σημαίνει ότι δημιουργούμε καινούριε θέσει εργασία στην Ευρώπη. Το είπα και πριν και θέλω να το επαναλάβω. Θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η σημαντική γεωπολιτική θέση της Σιγκαπούρης για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση κλιματικών φαινομένων στην όλη περιοχή είναι ιδιαίτερα σημαντική για μας. Η Σιγκαπούρη θα μπορέσει να βοηθήσει ε, ε, μάλλον εμείς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε την Σιγκαπούρη στην εφαρμογή των πολιτικών αποφάσεων που έχει πάρει για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής γιατί έχουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία. Τέλος να ευχαριστήσω τους και οδησηγητές για τη βοήθειά τους, για τη συνεργασία τους και ελπίζω ότι αύριο θα μπορέσουμε με ευρία πλειοψηφία να ε, ψηφίσουμε και να εγκρίνουμε αυτό το πλαίσιο συνεργασίας με τη Σιγκαπούρη. Είναι επιτυχία και επίτευγμα για όλους μας, ε, καθώς επίσης και ε, σημαντική πηγή σταθερότητας και θέσεων απασχόλησης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ήθελα ε, να τονίσω ότι ε, πρέπει να μιλάτε μία φωνή. Τώρα η κυρία Μάλμστρομ, εξ ονόματο των Ομοσιών. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σα κυρίε και κύριοι βουλευτές. Να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές, τον κύριο Ντέβιν Μάρτιν και τον κύριο Λόπες Ιστουρίς Βουάιτ για τη δουλειά που έχετε κάνει και την καινή σας πορεία που μας έφερε σήμερα εδώ. Λίγα μέρη συμβολίζουν τα πλεονεκτήματα του εμπορίου και των επενδύσεων όσο η Σιγκαπούρη, η οποία έχει ε, επιδείξει ένα ανοιχτό πνεύμα, μια παγκοσμιοποίηση και έχει μεταμορφωθεί χωρίς φυσικούς πόρους σε μια της πιο πλούσιες χώρες στον κόσμο. Η Σιγκαπούρη έχει γίνει υπόδειγμα οικονομικού μετασχηματισμού και χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς το εμπόριο επενδύσεις βιώσιμες ε, η βιώσιμη ανάπτυξη πάνε χέρι-χέρι. Και βεβαίως η ίδια αντίληψη ε, έχει ωφελήσει και εμά στο παρελθόν και πρέπει να μας καθοδηγεί και στο μέλλον. Ε, Στενή εταίρη, εδώ και δεκαετίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Σιγκαπούρη αποφάσισαν να επισφραγίσουν την ε, συνεργασία τους μέσω των τριών αυτών συμφωνιών. Η νέα αυτή συμφωνία θα θέσει το γενικότερο πλαίσιο της δημερούς συνεργασίας, πολιτικής συνεργασίας αλλά επίσης είμαστε και πολύ στενοί εταίροι εμπορίου και επενδύσεων. Είναι ο μεγαλύτερος μας εταίρος στην Ανατολική Ασία και στους 20 ε, κορυφαίους επενδυτές για αγαθά, στους 5 κορυφαίους ε, στις ε, επενδύσεις και από τους 10 κορυφαίους στο εμπόριο. Και έτσι θα αναπτυχθούν περισσότερο αυτοί οι δεσμοί. Τα ωφέλη είναι πολλά. Οι δασμοί στο διμερές εμπόριο θα καταργηθούν. Τα μη δασμολογικά φράγματα για ευρωπαϊκές εξαγωγές ε, επίσης ε, θα καταργηθούν. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες ε, δημόσιας προμήθειας θα βελτιωθεί. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και για τους ανθρώπους και στις δύο πλευρές. Επίσης υπάρχει ένα κεφάλαιο το οποίο αφορά το εμπόριο και την ανάπτυξη, τα δικαιώματα των εργαζομένων, το περιβάλλον, την βιοπικιλότητα, την οικολογική σήμανση, την εταιρική κοινωνική ευθύνη και πότε ένα σημαντικό ρόλο στις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών της Σιγκαπούρης. Η κύρωση και η συμμόρφωση με τις ε, συμβάσεις του ILO θα είναι από τα πρώτα σημεία τα οποία θα παρακολουθήσουμε και πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας ε, μέχρι να τεθεί ενισχύ συμφωνία. Και ήδη οι αρχές Σιγκαπούρης ε, προετοιμάζονται για την εφαρμογή των διατάξεων για την αηφόρο ανάπτυξη. Επίσης αυτά τα έχουμε διαπραγματευτεί σε συνδυασμό με μια συμφωνία για προστασία των επενδύσεων που έχει αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την οποία συνδιαμόρφωσε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σας ευχαριστώ. Το σύστημα αυτό αντιμετωπίζει τις ανησυχίες κοινωνίας των πολιτών για ασαφείς κανόνες, έλλειψη διαφάνειας, έλλειψη δυνατότητας ε, προσφυγής, ε, έλλειψη ανεξαρτησίας ε, των επιδιαιτητών. Οπότε, με βάση την διαπραγματευτική μας έντολη, σας παρουσιάζουμε μια συμφωνία η οποία καθιστά πιο αυστηρές αυτές τις προδιαγραφές για να μην υπάρξει κατάχρηση. Μια συμφωνία η οποία πλήρως σέβεται τα δικαιώματα των κυβερνήσεων να φέρουν νέα νομοθεσία για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος και άλλων δημοσίων αγαθών και δημιουργεί ένα πλήρως διάφανο σύστημα δικαστηρίων, κάτι το οποίο και ο Γενικός Αγγελέας ε, θεώρησε πλήρως συμβατό με τις συνθήκες ε, στην περίπτωση της συμφωνίας με τον Καναδά και θα μπορούσαμε έτσι να καλύψουμε και τις υφιστάμενες 3.000 εμπορικές συμφωνίες ε, παγκοσμίω. Και θα έχουμε έτσι μια εξέλιξη για να έχουμε και υποχρεώσεις των επενδυτών όπως ανέφερε ο κύριος Μάρτιν. Οπότε οι συμφωνίες αυτές είναι συμφωνίες που είναι πραγματικά η τελευταία λέξη των συμφωνιών αυτών και βεβαίως η Σιγκαπούρη είναι η καρδιά του εμπορίου της Νοτιοανατολικής Ασίας και θα αποτελέσει η συμφωνία αυτή ε, υπόδειγμα και για τους άλλους εταίρους. Και τέλος, ε, για την ε, Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών αποτελεί ένα περαιτέρω βήμα για εμά και τη Σιγκαπούρη αλλά και για ολόκληρη την περιοχή. Παρέχει μια βάση, όπω είπε ο εισηγητή, για αποτελεσματικέ διμερείς σχέσει με τη Σιγκαπούρη για ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου και για ενίσχυση τη συνεργασία σε πολλού τομεί, ε, Ανθρώπινα δικαιώματα, εργασιακά δικαιώματα, δικαιοσύνη, ασφάλεια, συνδεσιμότητα, διαπροσωπικές επαφές, ε, πληροφορική, πολιτιστικές ανταλλαγές, αλλά και απασχόληση και κοινωνικά. και θα μας επιτρέψει να εντείνουμε τις συνεργασίες τομείς όπως η ενέργεια, του περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή, η προστασία των φυσικών πόρων, έξυπνες πόλεις και μεταφορές. Και βεβαίως σε περίπτωση διαφωνιών θα συσταθεί μια διμερής επιτροπή υψηλού επίπεδου για την ορθή λειτουργία και εφαρμογή της ε, συμφωνίας αυτής και βεβαίως ε, θα προστατεύσουμε και τους στόχους της για την ε, περιφερειακή δυναμική. Η Σιγκαπούρη ε, μας έχει επιδείξει πως ε, είναι υπέρ της πολυμερούς προσέγγισης στην Νοτιοανατολική Ασία και εκτιμούμε ιδιαίτερο την συνεργασία μας και θα φροντίσουμε να γίνει ακόμα ισχυρότερη. Η συνεργασία με την Σιγκαπούρη για ζητήματα που αφορούν τον Αζίαν είναι πολύ επικοδομητική μέχρι στιγμή. Οπότε η συνεργασία των δύο μερών είναι βαθιά και ευρύτατη ήδη σήμερα και δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, οι δυνατότητε για ακόμα μεγαλύτερη συνεργασία είναι μεγάλε. Με βάση ένα κοινό όραμα, ένα πολυμερέ σύστημα που θα βασίζεται σε κανόνε Να ευχαριστήσω λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αναμένουμε την στήριξή σα στην αυριανή ψηφοφορία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Η αρχή της συζήτηση είναι πολλά υποσχόμενη, πολύ διαφορετικός ο τόνος από ό,τι στην προηγούμενη. Ο κύριος Κέλλη για το ΕΛΚ. Καταρχήν να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές. Πολύ καλή συνεργασία σε αυτό το θέμα και τους δυο εισηγητές θέλω να ευχαριστήσω. Καθυστέρησαν πολύ, αλλά ευτυχώς έχουμε φτάσει στο τέλος. Ελπίζω αύριο να ψηφίσουμε και να το εγκρίνουμε. Το εμπόριο ανάμεσα στην Καπούρ και την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει 55 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγέ για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 44 δισεκατομμύρια εξαγωγέ τη Σιγκαπούρη προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυξάνονται πολύ γρήγορα αυτά τα νούμερα, έτσι κι αλλιώ. Είναι πολύ καλή λοιπόν αυτή η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών. Συγχαίρω την κυρία Μάλστρομ για την πολύ καλή δουλειά τη. Ε, θα ωφεληθούν πολλοί κλάδοι. Ο πολιτικό κλάδο, για παράδειγμα, στην Ιρλανδία, όπω ξέρω. Αυτή η συμφωνία δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί για όλους, προς όφελος όλων. Με την απόσυρση των εμπορικών φραγμών, δασμολογικών και μη δασμολογικών, ε, κάνουμε ένα πολύ μεγάλο βήμα. Το πολυμερές δημοσιονομικό επενδυτικό δικαστήριο είναι μια πολύ καλή ιδέα. Και ε, μετά την αν συμφωνήσαμε τις συμφωνίες με τον Καναδά και την Ιαπωνία, σίγουρα θα πρέπει να συμφωνήσουμε και εδώ και μακάρι αύριο με λίγο Ιρλανδέζικο whisky να το γιορτάσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κέλλη. Θα μπορούσατε να σέβεστε λίγο το χρονικό όριο, το χρόνο που σας δίνουμε. Κυρία Μαρία Μόσκα. Επίτροπε, συνάδελφοι, λίγε εβδομάδε πριν την ψηφοφορία, ε, λίγε εβδομάδε μετά την ψηφοφορία του Κοινοβουλίου αυτού για τη συμφωνία με την Ιαπωνία, πάλι μιλάμε για τη σύναψη στρατηγική συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, του πολίτε τη, του εργαζομένου τη και τι επιχειρήσει τη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την ψηφοφορία ε, που δεν έγινε για τη συμφωνία με τι ΗΠΑ τώρα θέλει να γίνει πρωταγωνιστής στο διεθνές εμπορικό προσκήνιο. Η τρίτη οδός για το εμπόριο που θέλει να αντιμετωπίσει τον άκρατο ανταγωνισμό και τον ανεξέλεγκτο φιλελευθερισμό ποτέ δεν ήταν τόσο ελκυστική. Θα πρέπει να προαβάλουμε τις προδιαγραφές και τα πρότυπά μας σε διεθνές επίπεδο. Χάρη στις ρήτρες για την προστασία των εργαζομένων και των καταναλωτών, καθώς και του περιβάλλοντος, θα καταφέρουμε να προστατεύσουμε και τους πολίτε από τις παράπλευρες συνέπειε της παγκοσμιοποίησης. Για να αναφέρω μερικά, οι δεσμεύσει τη Σιγκαπούρη για την κύρωση των συμβάσεων του ILO, ε, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασία, για τον σεβασμό τη Συμφωνία ε, για το Κλίμα των Παρισίων, καθώ και την αναγνώριση των γεωγραφικών μα ενδείξεων, όπω η προστατευόμενη προέλευση και η προστατευόμενη καταγωγή. Εδώ θα, γεωγραφική ένδειξη, μάλλον. Εδώ θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια με την τέταρτη οικονομική δύναμη σε ανάπτυξη ε, και πώ θα φτάσουν τα προϊόντα στα σύνορά μα. Είναι μια σημαντική διέξοδο για να στηρίξουμε την απασχόληση και την ανάπτυξη ανάπτυξη. Η Σιγκαπούρη είναι μια ανοιχτή πόρτα για την ε, νοτιοανατολική Ασία, τι χώρε Αζιάν. Είναι η πιο δυναμική οικονομία του κόσμου. Είναι η 7 σε σημασία χώρα για τι εξαγωγέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. 30% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που έχουν παρουσία στην Σιγκαπούρη είναι μικρομεσαίε και οι εξαγωγέ έφεραν κέρδη 33 δι ευρώ στι επιχειρήσει μα. Η συμφωνία θα επιτρέψει να πολλαπλασιαστούν τα νούμερα αυτά και θα δημιουργήσει πολλαπλέ θέσει εργασία στην Ευρώπη χωρί κανένα κόστο. Η βιομηχανία στη Σιγκαπούρη είναι συμπληρωματική προ την Ευρωπαϊκή. Στον βιομηχανικό κλάδο αλλά και στη Γεωργία, δεν υπάρχει κανένα κομμάτι τη οικονομία μα που δεν θα ωφεληθεί από τη συνεργασία με τη Σιγκαπούρη. Σε σχέση με τα γεγονότα αυτά και τα αριθμητικά αυτά στοιχεία, δεν πρέπει να υπάρχουν αμφιβολίε. Οι συμφωνίε αυτέ είναι καθοριστική σημασία για του εργαζομένου τη Ευρώπη. Τα προϊόντα μα και τα αγαθά μα πολλούνται και ε, εκτιμώνται σε όλο τον κόσμο. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε στη συμφωνία αυτή, περιορίζοντα τι αρνητικέ συνέπειε τη παγκοσμιοποίηση. Ευχαριστούμε πολύ εκ μέρου του ECR, ο κ. Στάνοκ. Κύριε Πρόεδρε, η Συμφωνία Ελεύθερη Συνεργασία με τη Σιγκαπούρη είναι ένα ακόμα παράδειγμα τη ε, ε, επιτυχημένη εφαρμογή ε, το, το ανοίγματο των συνόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά την Ιαπωνία, για παράδειγμα, ανοίγουν αγορέ και άλλε αγορέ. Ε, η Βρετανία βρίσκεται 45 μέρε πριν την ε, αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αλλά να σας θυμίσω όλα αυτά τα οποία, τα ψευδή τα οποία είχαν υποσχεθεί οι υπέρμαχοι του Brexit από την, ε, για, για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τι υποσχόντουσαν, υποσχόντουσαν ότι η, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ενδιαφερόταν ούτε μπορούσε να συνάψει συμφωνίε που να ωφελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να όμως που βλέπουμε μια τέτοια συμφωνία ε, που έρχεται κατόπιν το συμφωνία με τον Καναδά, την Αυστραλία και, την, και και τη Νέα Ζηλανδία, ενώ οι συμφωνίε με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία είναι επίση πολύ προχωρημένε. Είναι προφανέ πλέον ότι μετά τι 29 Μαρτίου οι 27 χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν πολύ περισσότερε ευκαιρίε να κάνουν εμπόριο με τη Σιγκαπούρη από το Ηνωμένο Βασίλειο για τα επόμενα χρόνια. Ο κ. Τάισον, ε, επιχειρηματία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπέρ του Brexit, ε, έχει ήδη ξεκινήσει να χτίζει ένα εργοστάσιο ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη Σιγκαπούρη και μετέφερε την έδρα του από τη Βρετανία εκεί. Τι άλλο να πω, ευχαριστώ. Πρόεδρο. ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρου τη Άλντε, ο κ. Τερμόσεϊ Μπαλσέλς. Αγαπητέ κυρία Επιτροπέ, Κυρίε και κύριοι, να ξεκινήσω λέγοντα ότι η συνεργασία ανάμεσα στον David Μάρτκιν και τους κοιόδους ηγητές ήταν εξαιρετική και γι' αυτό το λόγο είχαμε ε, μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στην ψηφοφορία τη Επιτροπής ΙΝΤΑ. Επίση, να ευχαριστήσω τον πρέσβη τη Σιγκαπούρη και την κυβέρνηση Σιγκαπούρης για την ε, υπομονή του. Στηρίζω και την Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών και το Μηχανισμό προστασία Επενδύσεων. Είναι αμοιβαία ωφελό ε, αμοιβαίω ωφελή ε, συνεργασία και για τη Σιγκαπούρη και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι εταιρείε του. Οι διαπραγματεύσει ξεκίνησαν το 2009, Δεκέμβριο 2009. Σχεδόν 10 χρόνια μετά βρισκόμαστε στο τέλο του δρόμου αυτού. Ε, είναι ο, ο μεγαλύτερος ε, εταίρος μας στην περιοχή. Ε, πάνω από 10.000 ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν τα περιφερειακά τους γραφεία στην Καπούρη και δρούν σε ένα αξιόπιστο επενδυτικό περιβάλλον. Είναι επίσης ε, κόμβος ε, για όλη την Ασία Σιγκαπούρη, μεταφορικός και εμπορικός. Η συμφωνία αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει μοντέλο και για τις άλλες ασιατικές χώρες. Είναι η πρώτη σε αυτή την περιοχή που υπογράφουμε. Ε, η Συμφωνία Προστασίας των Επενδύσεων αντικαθιστά 13 διμερείς αντίστοιχες συμφωνίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μεταξύ κρατών μελών και τη Σιγκαπούρης. Αύριο Ελπίζω ότι θα υπερψηφίσουμε αυτό, αυτή την, αυτό το νέο, μοντέρνο σύστημα προστασίας επενδύσεων που θα μας βοηθήσει να εξασφαλίσουμε τους θεμητούς στόχους της εμπορικής μας πολιτικής δίνοντας ε, ε, ασφάλεια και προστατεύοντας το περιβάλλον. Επίσης, ε, η συμφωνία αυτή ορίζει μια μεταχείριση των εταιριών χωρίς διακρίσεις ε, και ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο. Θα ήθελα τέλος να αναγνωρίσω και να ευχαριστήσω την κυρία Μάλστρομ για τις προσπάθειές της. Ε, μας βοήθησε πάρα πολύ σε πλήρη διαφάνεια. Η ανάπτυξη στην Ευρώπη έρχεται με το εμπόριο, κυρίε και κύριοι, όχι με μεγαλύτερα κρατικά χρέη. Με τον Brexit και τον Τραμπ ο, η πολυμερής προσέγγιση κινδυνεύει. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Τώρα, αξιόνοματος ε, της ε, Γκουε, η κυρία Μαρή Κύριε Πρόεδρε, έχω τρεις σοβαρές επιφυλάξεις ε, για αυτήν τη συμφωνία. Περιλαμβάνεται πάλι μια παραγράφος για το ISDS, δηλαδή κάποιο διαιτητικό δικαστήριο για τους επενδυτές. Αυτό είναι κατ' ουσίαν. Γνωρίζουμε πως εδώ πέρα έχουν δικούς τους κανόνες ε, οι επιχειρήσεις και μπορούν να σέρνουν τα κράτη ενώπιον αυτού του δικαστηρίου και να πληρώνει ο φορολογούμενος. Εδώ πέρα υπονομεύεται το κράτος δικαίου και η δημοκρατία. Δεύτερον, η σύμβαση προσφέρει αποκλειστικά δικαιώματα σε επενδυτές, αλλά δεν υπάρχουν κανόνες υποχρεωτικοί για την υλοποίηση των διατάξεων περιφορίας. Εδώ πέρα λοιπόν θα υποφέρουν άνθρωποι, ζώα και περιβάλλον. Τρίτον, υπάρχει ρητά η δυνατότητα σε ξένους επενδυτές να αγοράσουν κρατικά ομόλογα και σε καιρούς κρίσης μπορούν να προχωρήσουν σε να μπλοκάρουν, συγχωρείτε, αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους το Κοινοβούλιο και οι Κομισιόν εδώ πέρα υπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα πολυεθνικών επενδυτών και τα βάζουν πάνω από το συμφέρον των πολιτών. Είναι απαράδεκτο. Σχεδόν μισό εκατομμύριο άνθρωποι την προηγούμενη εβδομάδα υπέγραψαν μια αίτηση κατά του ISDS ακριβώς για να σταματήσουν τέτοιες συμβάσεις. Σταματήστε λοιπόν το ISDS, σταματήστε αυτήν την εμπορική συνθήκη και σταματήστε την ταξική δικαιοσύνη για τις πολυεθνικές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα για τους πράσινους ο κύριος Μπιουτικόφερ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, το καλό πράγμα αργεί να γίνει, λέμε, στην ε, Γερμανία. Και βεβαίως άργησε πολύ. Και πρέπει να πω ότι ήταν πολύ υπομονετική η Σιγκαπούρη και την συγχαίρω ακριβώς για το τι βοήθησαν στον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Αζίαν. Η συμφωνία δείχνει ότι η Ευρώπη επιθυμεί την ενισχυμένη συνεργασία με τον Αζίαν για το συμφέρον μας και για τις αξίες μας. Χρειαζόμαστε στρατηγικές εταιρικές σχέσεις και χρειαζόμαστε μια τέτοια σχέση με τον Αζίαν για να προωθήσουμε την ασφάλεια και την ανάπτυξη στην περιοχή του Ινδικού και του Ειρηνικού ωκεανού και θέλουμε και πολυμερή συνεργασία και τέλος θέλουμε την πλήρη εφαρμογή των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την ελευθερία του συνέρχεστε μέχρι την κατάρριξη θανατικής ποινής. Αλλά επίσης πρέπει να θέσω ένα πρόβλημα και το λέω στα αγγλικά για να γίνει αντιληπτό και στην Σιγκαπούρη. Τα ομόλογα, δεν, τα κρατικά ομόλογα δεν θα πρέπει να καλύπτονται από τις συμφωνίες προστασίας των επενδυτών. Από την κρίση του 2007 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγκεκριμένες διαδικασίες για την αναδιάρθρωση χρέους σε περίπτωση χρεοκοπίας. Εδώ πέρα λοιπόν δημιουργείται ένα παραθυράκι με τη Συμφωνία της Σιγκαπούρης, όπως λέει και η Handelsblatt σήμερα, η συμφωνία αυτή αυξάνει το κατόφλι για την συνένεση των πενητών σε περίπτωση αναδιάρθρωσης χρέους σε σχέση με το επίπεδο που ισχύει αλλιώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι επενδυτές ε, που λειτουργούν με βάση αυτήν την συμφωνία έχουν προνόμια σχέση με άλλους επενδυτές και αυτό είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό απαιτούμε η συμφωνία αυτή να μην ψηφιστεί αύριο μέχρι να καταργηθεί το περάρτημα 4 για το δημόσιο χρέος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα μιλάτε χωρίς να σας δώσω το λόγο. Συνάδελφε, στο έδρανο 39. Σας παρακαλώ. Ωραία. Εκ μέρους του FTD, κυρία Μπαγκίν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, δεν μπορούμε να παραχωρήσουμε στις πολυεθνικές να κάνουν τη δουλειά των κρατών. Σε αυτό το κοινοβούλιο φαίνεται ότι όλοι συμμετέχουμε τον ίδιο τρόπο, αλλά και εσείς ε, εκπροσωπείτε με τον ίδιο τρόπο τους πολίτες, υποτίθεται. Δεν μπορείτε λοιπόν να βάλετε αποφάσεις σε αυτή τη σύνοδο χωρίς να είναι πραγματικά ανεξάρτητες. Δεν μπορεί να ψηφίζετε υπέρ μια συμφωνία για επενδύσεις με τη Σιγκαπούρη. Και είναι ακόμη χειρότερη η συμφωνία αυτή από τη ΣΕΤΑ. Οι πολυεθνικέ ουσιαστικά θα έχουν υποχείριο τις χώρες μας ε, τι κυβερνήσει, τι περιφέρειε, του αρχέ τη τοπική αυτοδιοίκηση θα μπορούν από ε, δικαστήρια επίλυση διαφορών επενδυτών κρατών να διαλυθούν τα κράτη, να ε, είναι θύματα των επενδυτών. Εγώ πιστεύω στο παγκόσμιο εμπόριο και πάντοτε το υποστηρίζω όταν μιλάμε για συγκεκριμένα κέρδη και ωφέλη για τι επιχειρήσει μα. Δεν μιλάμε μόνο για εμπόριο. Μιλάμε για συμφωνίε άλλου είδου και πρέπει να γίνει μια σαφή διάκριση. Υπάρχει συμφωνία για τι επενδύσει που θα επιτρέψει τι πολυεθνικέ να αποδηγετήσουν ουσιαστικά τα κράτη, αλλά υπάρχει και το θέμα των συναλλαγών, που αφορά μόνο τι εξαγωγέ και τι εισαγωγέ. Αυτή η διάσταση εισαγωγών-εξαγωγών είναι σίγουρα θετική για την ε, οικονομία μα. Θα μα επιτρέψει να αναπτυχθούμε σε μια νέα αγορά που θα εκμεταλλευτεί και την ανάπτυξη τη Αυστρία. τη Ασία, συγγνώμη. Εδώ όμω δεν χρειαζόμαστε μια τέτοια συμφωνία. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι οι διαπραγματεύσει αυτέ ε, εκπονήθηκαν με έλλειψη διαφάνεια και να πω ότι η Επιτροπή ενημέρωσε το Κοινοβούλιο μόνα για πράγματα που ήδη ήταν τελεσμένα γεγονότα και για το θέμα των γεωγραφικών ενδείξεων κυρίω. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θα κοιτάξουμε με ιδιαίτερη προφυλακτικότητα το πώ θα αντιδράσουμε στην ψήφιση αυτή τη συμφωνία. Και υπάρχει και το θέμα των επενδύσεων. Η συμφωνία για, την, ε, για τι επενδύσει περιέχει αυτή τη ρήτρα για την περιβόητη επίλυση των διαφορών και το σχετικό όργανο δικαστήριο. Είχαμε αντιταχθεί ε, έντονα και σφοδρά και στην ανάλογη διάταξη στη Συμφωνία ΣΕΤΑ και γι' αυτό μα έχουν ψηφίσει πολίτε. Για να καταψηφίζουμε τέτοιες είδου ιδέε. Ευχαριστούμε και τώρα ε, για την ΕΝΕΦ e ο κύριος Ζαμέ. Η κυρία Ζαμέ. Πρόεδρε, συνάδελφοι, εδώ το εμπόριο σίγουρα δεν ε, έχει δεν έχει την απαραίτητη ενέργεια, αλλά αυτό είναι το κρέντο, το πιστεύω των ε, γραφειοκρατών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταργώντα τα σύνορα, η συμφωνία με τη Σιγκαπούρη θα μα κάνει αποθήκη και ε, σταυροδρόμι του παγκόσμιου εμπορίου και θα προσθεθεί η συμφωνία αυτή σε όλε τι υπόλοιπε. Ανοίγουμε διάπλετα τι πόρτε μα στα εμπορεύματα τη Ασία, του Ειρηνικού, τη Νότια Αμερική. Κάτι που σίγουρα θα θέσει φιβόρο τη δική μα την οικονομία. Η συμφωνία αυτή μάλιστα είναι άκρο επικίνδυνη για του Γάλλου καταναλωτέ και του Ευρωπαίου καταναλωτέ. Γιατί η Σιγκαπούρη δεν αναγνωρίζει ένα μεγάλο μέρο των γεωγραφικών μα ενδείξεων. Ε, και των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Σε ό,τι αφορά τι ευρωπαϊκέ αξίε, να μην τι αναφέρω καν. Θα ήταν ε, κάτι που εκεί συστηματικά και επανειλημμένω ε, θα άρχιζαν τα συμφέροντα των πολυεθνικών. Η, ελευθερία, η ελευθεροτυπία, τα δικαιώματα των ανθρώπων, οι γκρίζε ζώνε των φορολογικών παραδείσων. Τίποτα από αυτά δεν ενοχλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το εμπόριο. Πάνω από όλα το εμπόριο, αυτή η παγκόσμια επιδημία. Μόνο που ούτε η Γαλλία, Ούτε η Ευρώπη δεν επωφελούνται από αυτέ τι συναλλαγέ των πολυεθνικών. Οι πολυεθνικέ επωφελούνται σίγουρα. Πάντω, αυτέ οι, οι άκρατε φιλελεύθερε ε, πολιτικέ είναι ουσιαστικά κοροϊδία τη οποία δεν θέλουν άλλο οι λαοί. Θέλουν η παραγωγή να επιστρέψει στην επικράτειά του. Τα προϊόντα να πηγαίνουν στι αγορέ που μπορούν να τα αγοράζουν εκείνη απευθεία και να τα βάζουν στο πιάτο του. Αντιτασσόμεστα σε αυτή τη συμφωνία με αυτή την πολιτική παγκοσμιοποίηση των αγαθών Ευρωπαίων των μακάριων Ευρωπαίων. Αυτό που θα εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα μπορέσει να το αποδεχτεί και να το καταπιεί ο λαό. Σα ευχαριστούμε και τώρα να περάσουμε στην ε, κυρία Κβίστφουντ Ρόβολ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα περιοριστώ σε κάποια σημεία μόνο. Πρώτον, ε, είναι η η πρώτη συμφωνία που έρχεται μετά την απόφαση του ΔΕΚ για την αποκλειστική ή μεικτή αρμοδιότητα για τέτοιες συμφωνίες. Οπότε είναι μια σύγχρονη ε, συμφωνία αυτή την οποία θα ψηφίσουμε. Δύο σημεία τώρα. Το πρώτο κομμάτι της ε, συμφωνίας αυτής ε, για τις ε, συμβάσεις του ILO. Η Σιγκαπούρη έχει δεσμευτεί γραπτός ότι θα τις κυρώσει. Ε, μα αυτό είναι αυτό που θέλουμε. Νομίζω ότι τελικά ε, είναι κάτι το οποίο είναι μια νίκη για εμάς και για την κυρία Επίτροπο για την προστασία των επενδύσεων. Έχουμε ένα διμερές δικαστήριο στο οποίο συμφωνήσαμε. Αυτό το οποίο δηλαδή ζητάμε εδώ και χρόνια σε αυτό το κοινοβούλιο είναι κάτι το οποίο πλέον έχει αναγνωριστεί γραπτός. Και αυτό θετικό για εμάς. Η Σιγκαπούρη θα μας ανοίξει την πόρτα για τις άλλες χώρες ε, του Αζίαν και αυτό θα το υπερψηφίσει ε, το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε τώρα στην κυρία Γκρας Βαντερ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, η Κομισιόν μας λέει συνεχώς ότι θα έχουμε εμπόριο για όλους, αλλά πάλι δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Έχουμε μια ριζοσπαστική πολιτική της αγοράς, από την οποία κερδίζουν μόνο μεγάλες εταιρείε. Αηφορία, δικαιώματα εργαζομένων και περιβαλλοντικές προδιαγραφές περνάνε σε δεύτερη μοίρα, να μην πω ότι αγνοούνται τελώ. Η Σιγκαπούρη δεν έχει κυρώσει τις 8 βασικές συμβάσεις του ILO. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει δυνατότητα κυρώσεων. Όμως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο κείμενο και το ICS βεβαίως ε, είναι κάποια βελτίωση, αλλά το βασικό πρόβλημα δεν έχει παραμεριστεί. Οι ξένοι επενδυτές εξακολουθούν να έχουν προνομιούχο θέση ε, και ξεπερνούν τα εθνικά δικαστήρια. Δεν είναι αυτό εμπόριο με βάση τους ε, κανόνες. Γι' αυτό θα καταψηφίσω και την εμπορική συμφωνία και την συμφωνία προστασίας των επενδύσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάνν Ζάχραντιλ. Ευχαριστώ. Είναι η τρίτη μου θητεία σε αυτό το κοινοβούλιο. Και θυμάμαι πόσο κόπο χρειαστήκαμε και πόσο χρόνο χρειαστήκαμε να φτάσουμε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Ήδη είχαμε ξεκινήσει από την προηγούμενη θητεία και μόλις τώρα ολοκληρώνουμε τις εργασίες μας. Η Σιγκαπούρη είναι κόμβος για την Νοτιοανατολική Ασία και συνολικά για την Ασία. Η απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου διευρύνεται μετά τη συμφωνία με την Ιαπωνία στη συγκεκριμένη περιοχή. Και ετοιμάζουμε και άλλη μια παρόμοια συμφωνία με το Βιετνάμ. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε πριν τελειώσει η θητεία μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σάκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επιτρόπε, κυρίες και κύριοι. Τα αγαθά ανταλλάσσονται εδώ και αιώνες και σε μεγάλες αποστάσεις όσο είχαμε τρόπο να τα μεταφέρουμε. Τώρα όλο και περισσότερο εξαιτία τη ψηφιοποίηση και οι υπηρεσίε μπορούν να προσφερθούν. Ένας μεταφραστής από την Ασία μπορεί να μεταφράσει ένα βιβλίο το οποίο έχει εκδοθεί εδώ, για παράδειγμα. Οπότε εμείς δεν δημιουργούμε εμπόριο. Αυτό που κάνουμε και πρέπει να κάνουμε είναι να διασφαλίζουμε ότι οι κανόνες που το διέπουν ε, είναι προβλέψιμοι και δίκαιοι. Θέλουμε υψηλότερε προδιαγραφέ και ε, να ωφελούμαστε όλοι. οι πρόεδροι Τσι και Τραμπ ε, δείχνουν τι μπορεί να προκληθεί από την έλλειψη κανόνων. Και είναι λίγο ηρωνικό το ότι επικρίνεται αυστηρά όχι τόσο το εμπόριο με την Κίνα για παράδειγμα αλλά οι κανόνες εμπορίου που θέλουμε εμεί να επιβάλλουμε μέσω των συμφωνιών. Οπότε χαίρομαι αυτούς που δείχνουν ότι είναι ηγέτες και τους εταίρους μας Σιγκαπούρη με τους οποίους διαπραγματευόμαστε εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Η Σιγκαπούρη είναι ένας μοντέρνος μίζων κόμπος στην περιοχή και ισχυρός μας εταίρος στην Νοτιοανατολική Ασία. Αλλά αυτή η συμφωνία δεν θα καταστήσει Σιγκαπούρενους Ευρωπαίους, ούτε και εμείς θα τους αντιγράψουμε. Όπως πάντα είμαστε υπεύθυνοι εμείς για την νομοθέτηση των δικών μας κοινωνιών. Και χαίρομαι που βλέπω ότι πείσαμε τη Σιγκαπούρη να αντικαταστήσει τις 13 πεπαλαιωμένες πλέον διμερείς συμφωνίες επενδύσεων ε, που έχει με κράτη-μέλη ε, και να ε, συμφωνήσει με την δημιουργία του καινούριου μηχανισμού προστασίας επενδύσεων, ο οποίος περιλαμβάνει ένα πρώτο βάθμιο δικαστήριο και δεύτερο βάθμιο δικαστήριο. Αυτοί που δεν συμφωνούν με την ISDS, με το μηχανισμό επίλυσης διαφορών, ε, θα πρέπει να είναι χαρούμενοι με αυτό το μοντέλο. Σε μια εποχή που προστατευτισμός, ο λαϊκισμός, ο εθνικισμός δείχνουν άνοδο, είναι σημαντικό να δώσουμε το χέρι στους εταίρους μας στο πλαίσιο τέτοιων συμφωνιών που βασίζονται σε κανόνες δίκαιους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κ. Μορέλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε. Οι συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών ε, ε, διαδέχονται μια την άλλη και μοιάζουν. Ε, σε επιτάχυνση, σχεδόν σε φρενήρια, μια και είμαστε στο τέλο τη θητεία, και μοιάζουν γιατί εξυπηρετούν κυρίω τα συμφέροντα όσων κατέχουν το κεφάλαιο ή των ιδιοκτητών των πολυεθνικών, ει βάρο των μισθωτών και των εργαζομένων. Τίποτα το καινούριο και σε αυτή τη συμφωνία με τη Σιγκαπούρη. Δεν υπάρχουν ε, περιορισμοί και απαιτήσει στα περιβαλλοντικά πρότυπα σε όσες ρήτρε ε, ουσιαστικά θα ευνοούν τις επιχειρήσεις ε, εις βάρος των κρατών, ούτε κάτι για τις επενδύσεις. Εδώ όμως θέλω να πω ότι οι ομόλογοι της Συγκαπούρης μας είπαν ότι έχουμε πολλές κοινέ αξίες με τις Ευρώπες. Μα δεν είναι καμιά ειρήνη και κοινοβουλευτική δημοκρατία, είναι ένα πολυτεχνικό καθεστώς η Συγκαπούρη. Επίσης, για μας πολύ σημαντικό είναι να σκεφτούμε την αντι, την αντίφαση αυτή. Είναι παγκόσμιο πρωταθλητή των φορολογικών παραδείσων, της αδιαφάνειας στα χρηματοοικονομικά. Από τη μια λοιπόν λέμε ότι θα ε, κυνηγάμε την ε, φοροδιαφυγή τη φοροαπάτη και από την άλλη με χαρά και σε τέτοια ψυχική εφορία θα εγκρίνουμε τέτοιε είδου συμφωνίε. Λέτε ότι είναι η καλύτερη συμφωνία που θα μπορούσαμε να έχουμε. Εγώ πιστεύω ότι ακόμα έχουμε πολύ δρόμο και πολύ κουπί. Ευχαριστώ. Ε, ο κύριος Ζαντό. Ε, εκ μέρους των Πρασίνων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε, ε, είπατε ότι είναι πολλά τα, οφ, ε, τα οικονομικά οι οικονομικέ δυνατότητε τη Σιγκαπούρη και ότι είναι υπόδειγμα. Όμω δεν μιλήσατε καθόλου για την ελευθεροτυπία και τη δημοκρατία. Αυτό δεν το αναφέρατε καν. Και δικαίω. Γιατί αυτή η συμφωνία επενδύσεων ουσιαστικά τι κάνει, ε, δεν ε, λαμβάνει καν υπόψη ότι δεν υπάρχει δημοκρατικό καθεστώ. Δεν βλέπετε ότι αναπτύσσονται οι εθνικισμοί, οι λαϊκισμοί. Δεν βλέπετε ότι όλα αυτά υποδαβλίζονται, ότι καλλιεργούνται από την ε, άρνηση τη εθνική κυριαρχία που οργανώνει οργανώνεται διαρκώ και την ενισχύεται ει βάρο των πολιτών. Το βλέπουν αυτό και ωφελείται τι πολυεθνικέ. Είναι δεκάδε οι πολυεθνικέ που έχουν έδρα στην ε, Σιγκαπούρη και θα επιτεθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την υγεία, το περιβάλλον, τι δημόσιε υπηρεσίε. Τώρα και για την αναδιάρθρωση του χρέου. Αυτό υπονομεύει τη δημοκρατία. Η Ευρώπη σημαίνει δημοκρατία. Η Ευρώπη θέλει του πολίτε τη. Δεν μπορεί να είναι για τι πολυεθνικέ. Επιτέλου, παρακαλώ, συνάδελφοι, απορρίψτε τη συμφωνία αυτή. Συλλήβδην. Δεν μπορούμε διαρκώ να υποστηρίζουμε τι δεν μπορούμε διαρκώ να υποστηρίζουμε του φορολογικού παραδείσου και τα πολυτερχία καθεστώτα. Αυτό υπονομεύει την δημοκρατία και καταστρέφει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε. Το μήνυμά σα ήταν σαφέ. Και τώρα... Earl of Dartmouth. Ναι, Πολύ καλό που κάποιο, και κάποιο άλλο ε, δείχνει τέτοιο πάθο. Η Σιγκαπούρη είναι μια επιτυχημένη ιστορία. Μια ιστορία επιτυχία. Έχει υψηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ από την ίδια τη Γερμανία. Αλλά η Σιγκαπούρη, επαναλαμβάνω, ε, δεν είναι, δεν είναι, επαναλαμβάνω, ένα τμήμα, τμήμα ενό μεγάλου εμπορικού ε, σχηματισμού. Και αυτοί που θέλουν η Βρετανία να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να το έχουν υπόψη τους. Και να απαντήσω στο προηγούμενο σχόλιο που έγινε. 45 χρόνια μετά την ένταξη της, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου υπογράφεται αυτή η συμφωνία. Πόσο πια θα μπορεί να καθυστερήσει κανένας. Αργά με γρήγορα βήματα εναλλάσσονται μεταξύ τους σαν χορό. Ε, αλλά αργό χορό. Ε, η θα γίνει αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Αλλά αυτό που δεν απαιτεί η συμφωνία είναι η ελευθερία διακίνησης ατόμων, προσώπων. Δηλαδή, το ελεύθερο εμπόριο ε, και η κυκλοφορία, ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων είναι πράγματα διαφορετικά. Ορίστε, αυτό λέγαμε κι εμείς ε, ε, για την Βρετανία. Δηλαδή, μπορούμε να καταργήσουμε τους δασμούς ε, χωρίς να έχουμε ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων. Αυτή τη στιγμή επαλευθερώνεται το εμπόριο στις υπηρεσίες. Ε, ταυτόχρονα όμως στη, η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να θέσει εμπόδια ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν ε, εξέλθει από, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δείχνει αυτή την κοινή λογική προς το Ηνωμένο Βασίλειο που δείχνει ήδη στη Σιγκαπούρη. Θα έρθει όμως μια μέρα που ο πρόεδρος του Συμφουλίου, ο κύριος Τάσκ, Τούσκ, θα βρει την θέση που του αξίζει στην κόλαση. Ο κύριος Τούσκ ε, ε, προσπαθεί να δηλητηριάσει την διαδικασία εξόδου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν θα το πετύχει. Οπότε συστήνω στι αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση να υπογράψουν μια παρόμοια συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, όπω αυτή που υπογράφουμε με τη Σιγκαπούρη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε μετά ε, ο κύριος, σας ευχαριστούμε για ο κύριος Λαντσίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούσαμε με μεγάλη προσοχή πόσο αποφελής και ε, θετική μπορεί να είναι η Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Σιγκαπούρη. Μου φαίνεται απίστευτο κάθε φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται μια εμπορική συμφωνία επενδύσεων με κάποιο άλλο μέρο ε, του κόσμου εκτό των σύνορων μα, πάντα είναι υποφελέ αμοιβαίω. Αυτή η συμφωνία ήταν αντικείμενο διαπραγματεύσεων σε μια εποχή που έχει ξεπεραστεί από τι εξελίξει τη πραγματικότητα. Στη Σιγκαπούρη, όπω φαίνεται από την πρόταση εμπορική συμφωνία, είναι ε, η κοιτίδα τη οικονομία και τη οικονομική ανάπτυξη τη Νοτιοανατολική Ασία. Όμω, συνάδελφοι, την οικονομική ανάπτυξη αυτή θα την ε, καρποθούν άλλοι που δεν είναι μέρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση με ευνοϊκέ εμπορικέ ρήτρε. Βλέπουμε ότι ε, η Σιγκαπούρη είναι τρίτη χώρα σε προέλευση παραπημένων προϊόντων στον κόσμο βάσει των μελετών. Καμία καταπολέμηση τη διαφθορά και η Ιταλική βιομηχανία είναι ένα από τα πρώτα θύματα των παραπημένων προϊόντων αυτών. Θα ανοίξουμε τι πόρτε σε προϊόντα τα οποία παράγονται με χαμηλό κόστο από τη Μαλαισία, την Κίνα και την ε, Ινδονησία και ε, στη Σιγκαπούρη απλώ φτάνουν για το τελευταίο στάδιο επεξεργασία του. Απομένουν πολλέ αμφιβολίε για τι γεωγραφικέ ενδείξει, την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. Το σύστημα που ισχύει στη Σιγκαπούρη δεν προβλέπει καν μητρό. Εδώ οι γεωγραφικέ ενδείξει ούτε καν αυτομάτω θα προστατεύονται. Οι Ευρωπαίοι ελεγκτέ θα πρέπει αυτονόμω να κινούν τη σχετική διαδικασία. Η Σιγκαπούρη είναι και κέντρο ε, χρηματοοικονομικών συναλλαγών με την αμοιβαία απελευθέρωση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Αυτό είναι ο βασικό σκοπό τη που θέλει να επιτρέψει να παρακάμπτονται ευρωπαϊκοί κανονισμοί για τα θέματα αυτά. Πολλέ ανεξάρτητε ε, ενώσει και οργανώσει ε, τοποθετούν τη Σιγκαπούρη σε, μια, σε έναν μαύρο κατάλογο φορολογικών παραδείσων παγκοσμίω ε, και με φορολογικό αποκλεισμό και με μεταφορά κερδών σε πολυεθνικές που έχουν έδρα στι ΗΠΑ. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον λόγο έχει ο κύριος Ντέιβιτ Μακάλιστερ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες μου και κύριοι, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση για την διάσταση της εξωτερικής πολιτικής, η οποία ήδη αναφέρθηκε ότι έχουμε ένα σύστημα που αναπτύχθηκε εδώ και δεκαετίες, ένα σύστημα πολυμερές παγκοσμίου εμπορίου το οποίο απειλείται και αμφισβητεί τις εταιρικές μας σχέσεις και προσπαθούν κάποιοι με προστατευτισμό να υπαναχωρήσουν από τα συμφωνηθέντα. Γι' αυτό λοιπόν η συμφωνία αυτή έρχεται την κατάλληλη στιγμή. Πηγαίνει πέρα από το καθαρά οικονομικό σκέλος, είναι ένα σημαντικό μήνυμα προς τους εταίρους μας ότι θέλουμε ένα πολυμερές σύστημα με κανόνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο έχει ο κύριος Γιώχιμ Σούστερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε περήφανοι ε, για το ότι δεν θέλουμε απλά ελεύθερο εμπόριο, αλλά με βάση τις αξίες. Και οπωσδήποτε αυτό σημαίνει ότι εμείς ε, και οι εταίροι μας έχουμε Κάποιε ελάχιστε προδιαγραφέ για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Γι' αυτό αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην κύρωση των συμβάσεων του ILO, του Διεθνού Γραφείου Εργασία. Η Σιγκαπούρη αρνείται να το κάνει αυτό ο υπουργό ε, Εμπορίου ε, από ό,τι φαίνεται έχει μια ιδιαίτερος εχθρική στάση. Αντί για συγκεκριμένα ε, χρονοδιαγράμματα, η επιστολή που μας απέθυναν περιέχει κάποιες γενικολογίες. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποια ελάχιστα δικαιώματα για τους εργαζόμενους, όχι μόνο για να προστατευτούν οι εργαζόμενοι εκεί πέρα. Το θέμα είναι να μην υπάρχει μισθολογικό ντάμπινγκ ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Είναι και ζήτημα αξιοπιστίας. Ε, δηλαδή, αν μιλάμε σοβαρά για εμπόριο που βασίζεται σε αξίες, πρέπει να απορρίψουμε αυτή τη συμφωνία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον λόγο έχει ο κύριος Μπιλ σας ευχαριστώ. Πόσο χαίρομαι που σας συναρπάζει μια εμπορική συμφωνία με μια δυναμική χώρα ε, νησιωτική με χαμηλούς φόρους. Συναρπαστικό και σας έχω νέα. Υπάρχει και άλλη μια τέτοια χώρα πολύ πιο κοντά ε, με την οποία μπορείτε να κάνετε μια συμφωνία όταν ξυπνήσετε βεβαίως. Βεβαίως όταν θα φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο η Σιγκαπούρη θα ε, μάλλον έχει ήδη πει ότι θέλει να κάνει συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο γιατί είμαστε δυναμικές ε, οικονομίες ε, που κινούμαστε γρήγορα δεν καθυστερούμε 10 χρόνια και μέχρι να σκόσουμε το ένα πόδι έχει βρωμίσει το άλλο λοιπόν μιλάμε για το εμπόριο μιλάμε για το πως θα γίνουμε πλουσιότεροι και θα εμπορευόμαστε προϊόντα και αγαθά. Δεν προσπαθούμε να επιβάλλουμε κανόνες ο ένας τον άλλον και να περνάει μια δεκαετία. Αναμένω λοιπόν τα ίδια συναρπαστικά να ζήσουμε και με το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα σας αρέσει πολύ. Ευχαριστώ. Ο κ. Κολομπιέ. Η σύναψη συμφωνία με τη Σιγκαπούρη ε, είναι σαν να βοηθάμε την Κίνα. Ε, το 75% των κατοίκων Σιγκαπούρης είναι Κινέζοι, οπότε ε, είναι η προφυλακή της Κίνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι, εξ, οι εξαγωγές της Σιγκαπούρης σε μεγάλο βαθμό είναι κινέζικα προϊόντα, τα οποία έχουν προηγουμένως εισαχθεί από την Κίνα. Η οικονομία της αγοράς δεν είναι κακό ως ε, έννοια, αλλά ε, το σημαντικό είναι να αποφύγουμε θανατηφόρες ανισορροπίες που μπορούν να καταστρέψουν τις οικονομίες μας. Εκεί δεν έχουν τις προδιαγραφές που έχουμε εμείς, ούτε τους κανόνες που έχουμε εμείς. Πολύ δε περισσότερο που το τραπεζικό του σύστημα είναι αδιαφανές. Αυτά μας δημιουργούν ανησυχίες. Οπότε, σας καλούμε να απορρίψετε αυτή τη συμφωνία, προκειμένου να προστατεύσουμε οικονομικά την Ευρώπη και ιδιαίτερως τη Γαλλία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος... Α, ναι, ο λόγος του κύριο Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να συγχαρώ τους εισηγητές. Ήδη υπογραμμίστηκε η στρατηγική σημασία της συμφωνίας αυτής με τη Σιγκαπούρη. Είναι ο πιο σημαντικός εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Νοτιοανατολική Ασία και τρίτος εξαγωγέας μετά την Κίνα και την Ιαπωνία από αυτή την περιοχή. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ακόμα περισσότερο την προσέγγιση ε, ενός ε, ελεύθερου εμπορίου δίκαιου και βασισμένου σε κανόνες. Οι συμφωνίες αυτές θα μπορούσαν να είχαν υπογραφεί πιο νωρίς, αυτό είναι αλήθεια, αλλά όπως είπε η κυρία Μάλστρομ, πολύ συχνά τον καιρό τη παγκόσμιοποίηση. δεν γίνεται λόγο μόνο για εισαγωγέ και εξαγωγέ, αλλά για πολύ περίπλοκε αλυσίδε παραγωγή με εισαγωγέ από διάφορα σημεία ε, τα οποία, ε, προϊόντα τα οποία συναρμολογούνται κάπου αλλού κλπ. Ευχαριστώ. Κέρτον Ντάρλινγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι στρατηγικό εταίρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση Σιγκαπούρη και πολύ σωστά προσπαθούμε να βαθύνουμε τη σχέση μα μαζί τη. Η συμφωνία αυτή θα αποτελέσει, οι συμφωνίε αυτέ θα αποτελέσουν μοντέλο για άλλε χώρε τη περιοχή. Οι εμπορικέ συμφωνίε όμω από μόνε του δεν χρησιμεύουν αν οι κανόνε οι οποίε διέπουν ωφελούν του λίγου και όχι του πολλού. Ε, η συμφωνία αυτή όμω έχει ένα πλαίσιο κανόνων. Ε, που όμως βασίστηκαν σε πολιτικές υποσχέσεις της τελευταίας στιγμής που μπορεί να μην υλοποιηθούν. Δεν θέλω να δοθούν περισσότερα προνόμια σε επιχειρήσεις, σε ανθρώπους όπως ο κύριος Γκουάμ, οι οποίοι βρίσκονται ενώπιν της δικαιοσύνης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κάσπαρη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Επιτέλους τελειώνει αυτή η διαδικασία και αύριο θα ψηφίσουμε αυτή τη συμφωνία. Είναι εδώ και χρόνια έτοιμη η συμφωνία. Ε, αποφασίσαμε όμως να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα με βάση αυτή τη συμφωνία ενώπιον του δικαστηρίου. Καμία άλλη συμφωνία δεν έχει εξεταστεί τόσο πολύ από το δικαστήριο όσο αυτή. Και επιτέλου ε, κάναμε με τη Σιγκαπούρη αυτό με το οποίο κάναμε με Καναδά και Ιαπωνία και θέλουμε να κάνουμε και με άλλε χώρε, δηλαδή κανόνε για το παγκόσμιο εμπόριο, έτσι ώστε να μην επικρατεί ο μεγαλύτερο και ισχυρότερο, όπω λένε κάποιοι συνάδελφοι, αλλά να υπάρχουν κανόνε και ένα σαφέ πλαίσιο. Γι' αυτό το ερώτημά μου προ του συναδέλφου που απορρίπτουν αυτή τη συμφωνία είναι τι θα προκύψει καλύτερο αν απορρίψουμε αυτή τη συμφωνία. Χάνουμε πολλές ευκαιρίες, αφήνουμε σε άλλους την αγορά, χάνουν τζίρο οι εργαζόμενοι μα. Ε, δεν βελτιώνουμε τίποτα εάν καταψηφίσουμε αυτή τη συμφωνία. Γι' αυτό παρακαλώ τους συναδέλφους να ξανασκεφτούν μέχρι αύριο τις τάσεις τους. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ και εγώ. Τον λόγο έχει ο κύριο Σίλβα Περέιρα. Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, το κοινοβούλιο μας πρέπει να εγκρίνει αμελητή τις τρεις σημαντικές αυτές συμφωνίες με τη Σιγκαπούρη που είναι ε, στο επιτάπητος για την οικονομία μας και για να δικαιωθεί η στατική σημασία της σχέσης με την Σιγκαπούρη. Ε, είναι σημαντικό για την πρόθεση των επενδύσεών μας, διότι είναι ακόμη ένα βήμα για την εκρίζωση των συστημάτων ιδιωτικού δικαίου και έτσι θα, περάσουν τρι, θα καταργηθούν τρει ε, διμερεί συμφωνίε που είναι επιχειωμένε. Επίση, η συμφωνία για την εμπορική θέμα γιατί διευκολύνει την εμπορική σχέση μα με ένα σημαντικό εταίρο στην Ανατολική Ασία, προωθεί την βιώσιμη ανάπτυξη και περιέχει συμβαστικέ μάλλον παραχωρήσει τη Σιγκαπούρη πολύ σημαντικέ για την κύρωση των ε, συμβάσεων του Διεθνού Οργανισμού Εργασία, του ILO. Επίση, ε, θα εγκρίνουμε ένα προοδευτικό ψήφισμα